Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, με την ιδιότητα της Προέδρου της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής, θα ήθελα να απευθύνω χαιρετισμό στα μέλη κατά την παρούσα κοινή συνεδρίαση ΔΕΚΑΜ και ΤΙΛΑΤ και ιδίω στο συμπρόεδρο αυτής της συνεδρίασης, τον κύριο Χαορεγγί, πρόεδρο της Αντιπροσωπείας Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρωπαϊκή Ένωση Λατινική Αμερική. Θα ήθελα επίση να καλούσω εγκάρδια την προσκεκλημένη μα, την κυρία Ιζαμπέλ Ντεμάλο Ντε Αλβαράδο, Αντιπρόεδρο και Υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Παναμά. Επίσης θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους εκπροσώπους διπλωματικών αποστολών και συγκεκριμένα την αυτού εξοχότητα τον κύριο Ντάριο Ερνέστο Σιρού Οκόα, πρέσβη της Δημοκρατίας του Παναμά, στου εκπροσώπου Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίω τον κύριο Πον, αναπληρωτή προϊστάμενο τη μονάδα για την Κεντρική Αμερική, το Μεξικό και την Καραϊβική τη Υπηρεσία Εξωτερική δράση. Η διερμηνία θα δυστυχώς δεν θα είναι μέχρι το τέλο τη ε, συνεδρίασης. Θα παρασχεθεί στα αγγλικά, ισπανικά, γερμανικά και ελληνικά ω συνεργητική γλώσσα και παθητική ιταλικά, γαλλικά, πορτογαλικά. Η συνεδρίαση θέλω να γνωρίζετε ότι μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου στον διαδικτυακό τόπο του Κοινοβουλίου. Το σχέδιο ημερήσια διάταξης σας έχει διανεμηθεί στα αγγλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, γαλλικά, γερμανικά και ελληνικά και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θα θεωρηθεί ότι η ημερήσια διάταξη έχει εγκριθεί. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια εκ μέρου τη ΔΕΚΑΜ. Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω την ευχαρίστησή μου για την επίσκεψη της αυτού εξοχότητας της κυρίας Ιζαμπέλ Ντεμάλο Ντεαλβαράδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κυρία, Αλβαράδο, η αντιπροσωπεία μας, <clears throat> είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει μια συνολική εικόνα της χώρας σας κατά την επίσκεψή της από τις 30 Μαρτίου ως την 1η Απριλίου του 2016. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θέσαμε επιτάπητος ένα μεγάλο φάσμα ζητημάτων από τις οικονομικές και πολιτικές πτυχές μέχρι την κοινωνική και νομική κατάσταση αλλά και τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αντιπροσωπεία μας πραγματοποίησε θετικές συζητήσεις με τους ομολόγους μας από την Εθνική Συνέλευση, τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, της επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας εντυπωσίασε την αντιπροσωπεία. Κατά τελευταία χρόνια η χώρα εξελίχθηκε σε μείζον σημασία παγκόσμιο εμπορικό κέντρο με πολύ ψηλά ποσοστά ανάπτυξης. Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε επίσης τη διόρυγα του Παναμά πριν από τα ιστορικά εγγένειά της στο άνοιγμά τη και την επέκτασή τη στι 26 Ιουνίου του 2016. Είχαμε επίση την ευκαιρία να ενημερωθούμε για την επιτυχή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παναμά στον τομέα της ασφάλειας κατά τη διάρκεια της επίσκεψή μας σε δύο συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργα στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΕΚΟΠΑ, το Κέντρο Αναμόρφωσης Ανηλίκων και το, Σοφρονιστικό Κέντρο Λανουεβα Χόγια. Κατά τη διάρκεια της επισκεψής μας, πολλοί από τους συνομιλητές μας τόνισαν τη σημασία της, μεγα... της γρήγορης επικύρωσης Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κεντρικής Αμερικής μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών έπραξα και έκανα κάθε δυνατή προσπάθεια για να πείσω τα κοινοβούλια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επισπεύσουν τη διαδικασία κύρωσης. Μέχρι σήμερα 20 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επικυρώσει τη συμφωνία και ελπίζουμε ότι και τα υπόλοιπα κοινοβούλια θα ακολουθήσουν σύντομα. Επιπλέον, κατά τι συναντήσει μα, συζητήσαμε τι προσπάθειε του Παναμά όσον αφορά στον αγώνα κατά τη φοροδιαφυγής και της νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε, και διαπιστώσαμε ότι στον τομέα τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε, ο Παναμά έχει συμμορφωθεί προ τα διεθνή πρότυπα, ενώ στον τομέα τη φοροδιαφυγής έχει συμμορφωθεί εν μέρη προ τα πρότυπα του ΩΣΑ. Δύο μέρε μετά την αναχώρηση αντιπροσωπεία μα από τον Παναμά, στι 3 Ιουλίου Απριλίου του 2016, μια ομάδα δημοσιογράφων από 76 χώρες, τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων, ξεκίνησε τη δημοσίευση εκθέσεων μετά από την διαρροή στοιχείων από την Τράπεζα Δεδομένων ενός δικηγορικού γραφείου του Παναμά, ε, το γραφείο Φωσέγκα. Η δημοσίευση αυτή προκάλεσε το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα σκάνδαλο όσον αφορά στην παγκόσμια αντιμετώπιση φορολογική απάτη, στην φοροδιαφυγή και την ομοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε. Συζητήσαμε επίση το θέμα στη συνεδρίαση της αντιπροσωπείας μας 21 Απριλίου του 2017. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να στήσει εξεταστική επιτροπή για τη διαρεύνηση των επανομαζόμενων εγγράφων του Παναμά, η οποία είχε στην, την καταστατική τη συνεδρίαση στι 12 Ιουλίου του 2016. Δεδομένου του τεράστιου φόρτου εργασία, η εντολή τη παρατάθηκε πρόσφατα μέχρι και τι 8 Δεκεμβρίου του 2017. Περιμένω λοιπόν με ανυπομονησία την ενημέρωσή σα σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν από τον Παναμά για την ενίσχυση τη καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και τη νομοποίησης εσόδων από παράνομε δραστηριότητε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Συμπρόεδρο, τον κύριο Χαουρεγγί. Ευχαριστώ πολύ Σοφία. Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω και να καλωσορίσω και την Αντιπρόεδρο του Παναμά, όπως επίσης και όσους εδώ εκπροσωπούν την κοινότητα της Κεντρικής και της Λατινικής Αμερικής, όλους τους φίλους συναδέλφους. Ξέρω πως έχει μια συνάντηση η Αντιπρόεδρος με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου στις 11. Μόλις έχει συναντηθεί με το ε, Συμβούλιο ε, σε μια συνεδρίαση που ε, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μάλιστα ήταν μια συνάντηση, ένα γεύμα εργασία, ένα πρωινό, στο οποίο συζήτησε πολύ ενδιαφέροντα θέματα με τα κράτη-μέλη. Θα περάσει βέβαια και από τη δική μα συνεδρίαση, όπου έχουμε τι αντιπροσωπείε για τη συνεργασία με τι χώρε Κεντρική Αμερική, Λατινική Αμερική, όπω επίση και του συναδέλφου από την Επιτροπή που έχουμε θεσπίσει για τη διερεύνηση του, θέμα, του θέματο των εγγράφων του Παναμά. Έχουμε λοιπόν πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μα. Να σα πω πω εδώ θέλουμε να συζητήσουμε τη διαφάνεια και όπως ε, ε, είπε και η κυρία Σακοράφα, να ζητήσουμε και για το θέμα των μεταρρυθμίσεων που έχει κάνει η κυβέρνηση σχετικά με το θέμα αυτό. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, κυρίες και κύριοι, μέλη του Προεδρείου, ε, αγαπητοί ευρωβουλευτές και ε, ε αγαπητοί συνάδελφοι από τις αντιπροπείες άλλων χωρών. Θα ήθελα να ξεκινήσω ε, εκφράζοντας πόσο λυπάται ο Παναμάς ε, για τα όσα συνέβησαν χθες στο Ηνωμένο Βασίλειο στην πρώτη επέτειο των γεγονότων των Βρυξελών, των νομοκρατικών επιθέσεων εκεί. Αυτό δείχνει πόσο εύθραυστοι είμαστε, πόσο ευάλωτοι και πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Ε, βεβαίω καταδικάζουμε τέτοιου είδου ε, βίαιε ναι. επιθέσει. Θα ήθελα να ξεκινήσω την παρέμβασή μου ευχαριστώντα ιδιαίτερα και με κάθε ειλικρίνεια τη αντιπροσωπεία ε, Eurolat και Eurocam για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συμμεριστούμε μαζί σας το νέο μας όραμα για τους βασικούς στόχους και ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν και οι δύο μας περιοχές. Ε, ξέρετε πως ε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για το ενδιαφέρον που έχετε δείξει για τη ε, χώρα μου και θα προσπαθήσω στο σύντομο χρόνο που έχω να μοιραστώ μαζί σας κάποια θέματα ε, που μας απασχολούν. Είναι ένας χώρος που είναι πολύ, πολύτιμος για τον Παναμά γιατί μας βοηθάει η δική σας, η συνεργασία μαζί σας να, μια και εκφράζετε την Ευρώπη, να εξηγήσουμε στη σημερινή συγκυρία περιφερεια, την περιφερειακή και τη διεθνή, τι ακριβώς κάνουμε στον Παναμά και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε μεταξύ τα δύο μπλοκ. Είναι ένα ε, σημείο χρονικό πολύ σημαντικό, γιατί αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις, αλλά παράλληλα και νέες ευκαιρίες. Και αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι γιατί εμεί από τον Νότο κοιτάμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το τι συμβαίνει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί για μας τους Λατινοαμερικάνους είναι μια δύναμη, είναι ένα μοντέλο, είναι αξίε τι οποίες μοιραζόμαστε και εμείς ε, σε επίπεδο ανθρωπινών δικαιωμάτων, δημοκρατίας. Είναι ένα μοντέλο το οποίο για μας είναι μοντέλο ε, περιφερειακής ενσωμάτωσης με εργαλεία για τη δημοκρατία, την ειρήνη, τη βιώσιμη ανάπτυξη που αποτελούν κομμάτια των προσδοκιών που έχουμε όχι μόνο για τη χώρα μα αλλά για την ευρύτερη περιοχή της Λατινική Αμερικής. Εμείς θεωρούμε πως η Λατινική Αμερική είναι ένας από τους πιο σημαντικούς συμμάχους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, επιτρέψτε μου να το εκφράσω, όχι μόνο γιατί έχουμε αυτέ τι κοινέ αξίε αλλά γιατί προσφέρουμε και ε, ευκαιρίες ε, αμφότεροι και να σας πω πως ε, οι πολυμερείς σχέσεις που έχουμε μας έχει βοηθήσει στο να εκφραστεί αυτή η φυσική συμμαχία μεταξύ μας. Έχουμε κάποιους μηχανισμούς που υπάρχουν που μας επιτρέπουν αυτή την προσέγγιση, αυτή την συστράτευση και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας σημαντικός παγκόσμιος παίκτη που καλό θα είναι να ενισχύσει σχέσεις που έχει με την Λατινική Αμερική και ε, το είπατε κι εσείς κυρία Πρόεδρε, Κάποιες χώρες έχουν ήδη κυρώσει αυτά τα ε, εργαλεία, αλλά αν μείνουν απλά λόγια σε ένα χαρτί, δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό που θέλουμε είναι αυτά τα εργαλεία να λάβουν σάρκα και οστά και να δημιουργήσουμε αυτή αυτούς τους ε, στενούς δεσμούς που είναι ευνοϊκοί για όλους μας. Και τις τελευταίες δύο δεκαετίες, δυόμιση δεκαετίες, εμείς αυτή τη στιγμή οικοδομήσαμε ένα πολύ πλούσιο και εκτιμένο μεταξύ των δύο περιφερειών μας σε πολλά στρατηγικά σημεία. Αλλά για να ανανεώσουμε, να αναζωπηρώσουμε αυτή τη ε, ε, συμμαχία, είναι επίγον να συμμορφωθούμε με τις νέες συστάσεις που αποφασίστηκαν στη σύνοδο μεταξύ μας το 2015. Θα πρέπει να ξαναβρούμε το δρόμο μας, να ξαναχαράξουμε πορεία έτσι ώστε να ε, συμμορφωθούμε με τους στόχους ε, της Agenda 2030 και με τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, όπως επίσης και τη Συμφωνία, τη Συνθήκη της Αντίσα Μπέμπα για την χρηματοδότηση, την αναπτυξιακή χρηματοδότηση. Και ξέρω πως εσείς έχετε πάρα πολλούς στόχους και πρέπει να σας πω πως από την Λατινική Αμερική, από την Καραϊβική, εμείς είμαστε σίγουροι πως αυτοί οι παγκόσμιοι στόχοι θα επιτευχθούν και μάλιστα θα ξεπεραστούν εάν συνεργαστούμε σε στενή ε, συμμαχία για να ε, χρησιμοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα, τα ανταγωνιστικά που προσφέρει και η μία και η άλλη περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει μία πορεία για να ανανεώσει με τη Χιλή και το Μεξικό τις συμφωνίες που έχει. Ξαναξεκίνησε διαπραγματεύσεις με το Μερκοσούρ και θα συμπληρώσουν αυτά τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με την Κολομβία, το Περού και τον Ισημερινό. Είναι λοιπόν επίγον να κλείσει η διαδικασία της κύρωσης της ε, ε, συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωση και Κεντρικής Αμερικής, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι πυλώνες που είναι ο διάλογος σε πολιτικό επίπεδο, η συνεργασία και η εμπορική συνεργασία. Εμείς είμαστε σίγουροι που στην επόμενη σύνοδο που θα γίνει στο Ελ Σαλβαδόρ θα έχουμε μια καταπληκτική ευκαιρία έτσι ώστε να αναζωπυρώσουμε αυτή αυτή τη φάση της στρατηγικής μας συμμαχίας και να γίνει μια συνάντηση μεταξύ των χωρών μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, μια και πρέπει να σας πω πως αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε την Προεδρία της ε, Ένωσης των χωρών της Κεντρικής Αμερικής και πιστεύω πως έχουμε μια ε, ευκαιρία να συνεργαστούμε σε πάρα πολλούς χώρους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μου αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει μια ηγετική θέση σε θέματα τα οποία ενδιαφέρουν ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από κάποιους μήνες, εμείς ήμασταν οι πρωταγωνιστές ε, στην, ε, στα εγγένεια μιας, ενός καταπληκτικού έργου που είναι η Νέα Διόρυγα του Παναμά. Ένα έργο μηχανικής καταπληκτικό και Πρέπει να σας πω πως ε, αυτή τη στιγμή πέρασε το χιλιοστό καράβι από ε, τα νέα τεχνικά έργα διασχίζοντας ολόκληρη τη διόργα και αυτό αποδεικνύει πόσο επιτυχημένο ήταν αυτό το έργο ε, στο οποίο πήραν μέρος πάρα πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες και αποτελεί ένα έργο πρόκληση το οποίο δείχνει ποιο είναι το δυναμικό μας και πόσο πολύ μπορούμε να προχωρήσουμε. Υπάρχει λοιπόν μια σύνδεση που προσφέρει ο Παναμάς που είναι που βασίζεται σε μια αναπτυσσόμενη στέρεα οικονομία που μας έκανε το δεύτερο πιο ανταγωνιστικό ε, κράτος της ε, περιοχής μας και είμαστε το κράτος με το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης. Και πρέπει να σας πω πως ο, ο κλάδος της, ε, των υπηρεσιών είναι τρίτα της οικονομίας μας και ε, είναι το 20% του ΑΕΠ και μάλιστα είναι αυτή η πτυχή της οικονομίας μας που μας επέτρεψε να ξεπεράσουμε τις αρνητικές διαστάσεις ε, της οικονομικής συγκυρίας σε διεθνές επίπεδο. Και είμαστε μια οικονομία η οποία ε, σέβεται και προωθεί το διεθνές δίκαιο, είναι διάφανη και έχει μία ε, απόλυτη δέσμευση με τα παγκόσμια πρότυπα για την χρηστή φορολογική και οικονομική ε, διακυβέρνηση. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να εμβαθύνουμε ε, στο θέμα αυτό και πρέπει να σας πω πως η κυβέρνησή μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει προσπαθήσει να ε, προσαρμοστεί στα πιο υψηλά επίπεδα και πρότυπα που επιβάλλει η Εθνική Συνεργασία και με ιδιαίτερη περηφάνεια μπορώ να σας πω ότι σήμερα οι δικές μας φορολογικές πολιτικές είναι στεναρές, ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα διεθνώς και ο πρόεδρος Βαρέλα που ήταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης στην προηγούμενη κυβέρνηση έχει υπογράψει αυτές τις συμφωνίες διπλής φορολόγησης ε, και πρέπει να σας πω πως αναγνωρίζω πως για κάποια τρία χρόνια ε, ο Παναμάς είχε ε, κατά κάποιο τρόπο ρίξει τους ρυθμούς του δυστυχώς πρέπει να το αναγνωρίσω αυτό όμως τώρα έχουμε ξανά πιάσει το ρυθμό πλεύσης. Αυτή τη στιγμή ενημερώνουμε τα μέτρα που έχουμε λάβει. Εμείς πριν από δυόμιση χρόνια αναλάβαμε ε, καθήκοντα και ο δικό χάρτης που έχουμε χαράξει είναι επιθετικός. Ο πρώτος στόχος που έχουμε είναι μέσα σε εννέα μήνες, δηλαδή χρόνο ρεκόρ, να βγούμε από τον ε, κατάλογο ε, των χωρών, ε, των ύποπτων των χωρών, να μας χαρακτηρίσω έτσι, και σύμφωνα με τα όσα έκανε ο πρόεδρος ε, Βαρέλα, υπογράψαμε όλους τους σχετικούς μηχανισμούς και πρέπει να σας πω ότι πλέον καταφέραμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Βέβαια, τα Panama Papers ήταν ένα τεράστιο χτύπημα για τη φήμη της χώρας μου και αυτή τη στιγμή ακολουθούμε έναν οδικό χάρτη, ο οποίος μας είχε επιτρέψει να ξεφύγουμε από το φαιό κατάλογο και να είμαστε αυτή τη στιγμή από τα κράτη τα οποία οποία κάνουν αυτομάτω ανταλλαγή πληροφοριών και όλα αυτά βεβαίω υπό την πίεση ε, να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν. Κάτι το οποίο επαναλαμβάνω κατακτήσαμε. Αυτή τη στιγμή ενισχύουμε την ανάπτυξη νέων προϊόντων και έχουμε ενισχύσει του θεσμού μα. Ξέρουμε σαφέστατα ποιε είναι οι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε και πρέπει να σα πω πω έχουμε ε, ε, εφαρμόσει επίση όλοι ή μάλλον έχουμε υιοθετήσει όλη την απαραίτητη νομοθεσία έτσι ώστε να ακολουθούμε εμεί. τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και να οικοδομήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο οτιδήποτε θα μας ε, επιτρέψει να ε, θέσουμε σε εφαρμογή όλες τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε και όλες τις συστάσεις που μας έγιναν. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με την πρώτη ανταλλαγή, ε, αυτό με την ανταλλαγή πληροφοριών τον Ιανουάριο του 2018 και αυτό δείχνει τι σημασία αποδίδει ο Παναμάς στο θέμα αυτό και εδώ έχω ε, το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Εσόδων του Παναμά που είναι εδώ για να σας περιγράψει τι προσπάθειες κάνουμε. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε την αυτόματη ανταλλαγή στοιχείων από το 2018 σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουμε υπογράψει. Και έχουμε αυτά τα reporting standards ε, του ΩΣΑ τα οποία ε, ακολουθούμε. Και πρέπει να σας πω ότι στη Γενική Γραμματεία του ΟΣΑ την περασμένη εβδομάδα καταθέσαμε τα εργαλεία που κυρώνουν ε, τη δική μας προσχώρηση στην Σύμβαση για την Διοικητική Αρρωγή, αμοιβαία αρρωγή σε φορολογικά θέματα. Και πρέπει να σας πω ότι θα ανταλλάσσουμε πλέον με πάνω από 100 χώρες τέτοιου είδους φορολογικές πληροφορίες. Αυτό κυρώθηκε και από την Γενική Συνέλευση, δηλαδή το Κοινοβούλιο μας και κατατέθηκε το εργαλείο αυτό την περασμένη εβδομάδα. Ε, προσαρμόσαμε το νομικό πλαίσιο που υποχρεώνει τις εταιρείε ε, στον ε, Παναμά να διατηρούν μητρώα, λογιστικά μητρώα και πληροφορίες για τις συναλλαγές που ασκούν. Και πρέπει να σας πω πως στα τέλη του μηνός θα εφαρμόσουμε και την διαδικασία αναθεώρησης που θα επιτρέψει να ξεφύγουμε από το χαρακτηρισμό που ε, δυστυχώς ε, έγινε ε, πρόσφατα, έτσι ώστε να μην είμαστε πλέον στον κατάλογο των χωρών που δεν συνεργάζονται. Και ζητάμε από τον ΩΣΑ να επιταχύνει την αξιολόγηση αυτή, έτσι ώστε να γίνουν κατανοητά τα πολύ σημαντικά βήματα που έκανε και πολύ γρήγορα βήματα που έκανε η χώρα μου, η για να ξεφύγει από αυτή την κατηγορία χωρών και να είμαστε σίγουροι πως η χώρα μας δεν είναι πλέον κομμάτι αυτών των ε, χωρών που δεν συνεργάζονται όπως ε, λέει η ομάδα των 20 ε, πιο αναπτυγμένων χωρών, η G20 και πρέπει να σας πω πως Είμαι εδώ και ζητώ από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μας στηρίξουν και να επαληθεύσετε κι εσείς ακριβώς τι βήματα ε, έκανε ο Παναμάς, γιατί είναι πολύ μεγάλη η πρόκληση αυτή. Δεν είμαστε πια φορολογικός παράδεισος. Τώρα, για την βάση, τη φορολογητέα βάση και τη μεταφορά κερδών, δηλαδή το BEPS, αν πούμε ε, τα αρχικά στα αγγλικά, να σας πω πώς θα αναθεωρήσουμε αυτές τις φορολογικές πρακτικές στις διάφορες δικαιοδοσίες που έχουμε και νομίζω ότι ε, και εκεί θα τα πάμε καλά και καταλαβαίνουμε πως θα πρέπει να είμαστε πάντα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να δείχνουμε και να αποδεικνύουμε τι αλλαγές έχουμε φέρει και έχουμε επιβάλει έτσι ώστε να είμαστε κι εμείς πάντα στην αιχμή του δόρατος ε, στα παγκόσμια πρότυπα. Και πρέπει να σας πω πως έχουμε μια σφαιρική στρατηγική ε, που εκτός από ε, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και νέες ευκαιρίες, εμείς τον Απρίλιο του 2016 δημιουργήσαμε, πρόεδρος δηλαδή Βαρέλα, μία επιτροπή με ε, ε, ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες έτσι ώστε να έχουμε συστάσεις για τη διαφάνεια της χρηματοσπιτικής μας ε, πλατφόρμας και για τις διεθνείς υπηρεσίες που προσφέρουμε και αυτή τη στιγμή έχουμε εντάξει αυτές τις συστάσεις στον οδικό χάρτη που προετοιμάσαμε για να μας οδηγήσει σε αυτή τη νέα εποχή. Και πρέπει να σας πω πως για το ξέπλυμα χρήματος και για τα παράνομα έσοδα είναι παγκόσμιο πρόβλημα και απαιτούν παγκόσμια λύση. Εμείς έχουμε οδικό χάρτη, θα ακολουθήσουμε τα όσα έχουμε εκεί, αλλά είναι μια μάχη υπέρ της οποίας έχουμε δεσμευθεί, αλλά χρειαζόμαστε να έχουμε μεταβατικές περιόδους, εύλογα χρονικά ε, διαστήματα έτσι ώστε να εφαρμόσουμε τις αλλαγές χωρίς τραύματα σε ε, τοπικό επίπεδο να μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Γιατί θα πρέπει να έχουμε αναλογικότητα με τα μέτρα που θα εφαρμόσουμε, το κόστος των μέτρων και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για μικρές χώρες όπως η δική μου οι εναλλακτικέ λύσει που έχουν οι χώρε μέσω εισοδήματο για να βρουν του πόρου ε, που θα του επιτρέψει τη βιώσιμη ανάπτυξη που είναι ο στόχο υπέρ του οποίου έχουμε όλοι δεσμευτεί. Με αυτά θα κλείσω. Θα κλείσω υπογραμμίζοντα τη δέσμευση τη χώρα μου να συνεχίσει να προχωράει ακολουθώντα την καλύτερη παράδοση του Παναμά, δηλαδή να βρει ε, κοινέ οδού που θα επιτρέψουν στον Παναμά να συνεργαστεί με την ε, διεθνή κοινότητα και τι προσπάθειε που γίνονται εκεί. εμεί θα σταθούμε δίπλα σας και θα καταφέρουμε κάποια ε, κοινά συμφέροντα που θα μας ευνοήσουν όλους. Αυτή είναι η δέσμευση που αναλαμβάνουμε εμείς και έναντι και ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με ολόκληρο τον πλανήτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να έρθω εδώ και να μοιραστώ μαζί σας σήμερα, παρόλο που καταλαβαίνετε ήταν πολύ σύντομο το διάστημα που είχαμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστούμε πολύ ε, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε λίγα, λίγο χρόνο στη διάθεσή μας έτσι ώστε να τεθούν ερωτήσεις και να έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε. Θα ήθελα να παρακαλέσω ε, η κάθε ε, παρέμβαση να μην ξεπεράσει το 1-1,5 λεπτό. Ε, ο κύριος Μάτο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Αποστολής, ζήτησε να είναι εδώ και θα είναι μαζί σας, γιατί εγώ ζητώ συγγνώμη, πρέπει να φύγω στις 10.30. επίσης, είναι, έχουν εγγραφεί η Ρενάτα Βέβερ, ο Εγνάθο Φαρίγια, και νομίζω ότι τέσσερις θα είναι στην αρχή ε, ή ε, παρεμβαίνοντας. Ένας τον Ευχαριστώ πολύ, Ραμόν. Κυρία Αντιπρόεδρε, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά λόγια που είπατε, αλλά ε, η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε κάποιες αμφιβολίες για την ταχύτητα με την οποία ε, θα προχωρήσουν τα πράγματα. Έχω και κάποιες ερωτήσεις. Ε, η ε, Διαρευνητική Επιτροπή, η οποία ξεκίνησε, αποχώρησε από τον Παναμά και εγώ θα ήθελα να ξέρω ακριβώς πώς προχώρησαν τα πράγματα, γιατί ε, ε, εμείς στην ε, δική μας Επιτροπή Ελέγχου των Panama Papers ακούσαμε πολλούς έγκριτους επιστήμονες οι οποίοι επίσης εξέφρασαν κάποιες αμφιβολίες. Δεύτερον, προετοιμάζεται κάποιο σύστημα πληροφορικής έτσι ώστε να προχωρήσετε στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Επίσης, τι γίνεται με τις, με τις εταιρείες οι οποίες είναι ε, ε, τι κάνετε ε, με αυτές, τι κάνετε όσον αφορά τους beneficial owners, τους τελικούς πραγματικούς ιδιοκτήτες. Έχετε κάνει κάτι, έχετε προχωρήσει σε αυτό. Νομίζω ότι πέρα από τα καλά λόγια τα οποία εκτιμούμε και πέρα από τις βαρύδουπες δηλώσεις θέλουμε να ξέρουμε στην ουσία τι γίνεται. Ευχαριστώ. Θα απαντήσει άμεσα ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ειλικρίνεια των ερωτήσεών σας και μας δίνετε τη δυνατότητα να πάμε πραγματικά στην ουσία του πράγματος. Ε, κοιτάξτε, ε, το Φόρο Global ε, ναι, ξεκίνησε μια fast track, γρήγορη διαδικασία αξιολόγηση, γιατί ε, είναι γεγονό ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διερευνηθούν και οι δικέ μα μεταρρυθμίσει. εγώ θα ήθελα να, μπορείτε, να, να, να, μπορούσατε να έρθετε, να δείτε από κοντά ότι πραγματικά είναι αυτά τα οποία δηλώνουμε και δεν τα δηλώνουμε απλώ έτσι για να πούμε μεγάλε κουβέντε. Όσον αφορά ε, την ε, Πολυμερή Επιτροπή, ε, η οποία επιτρέπει στον, στον Παναμά συγγνώμη, ανταλλαγή πληροφοριών. Πρέπει να σας πω ότι, όπως είπα και προηγούμενος, έχουμε εδώ και τον Γενικό Γραμματέα Εσόδων, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με το θέμα. Βεβαίως, έχουμε απόλυτη γνώση και επίγνωση ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και πολλά πρέπει να γίνουν εδώ. Κάνουμε ένα πρώτο βήμα και οπωσδήποτε θα πρέπει να ακολουθήσει άμεσα η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2018. Έχει επίγνωση η χώρα μου ότι η πρόκληση είναι μεγάλη ε, και ότι ο κίνδυνος είναι επίσης ε, ε, πάρα πολύ μεγάλος, κυρίως σε σχέση με το τι θα γίνει αν δεν καταφέρουμε να επιτύχουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά πρέπει να σας πω ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δυστυχώς ο χρόνος δεν μου επιτρέπει να μοιραστώ μαζί σας και να σας τα αναφέρω. Έχετε δίκιο ότι οι ανώνυμες εταιρείε οι οποίες έχουν καταγραφεί στον Παναμά, είναι εγγεγραμμένες δηλαδή στον Παναμά, αλλά δεν έχουν δραστηριότητα ε, στην χώρα ε, αποτελούν ένα πρόβλημα. Για αυτές ε, τις εταιρείες εμείς έχουμε εγκρίνει νομοθεσία η οποία δίνει τη δυνατότητα παροχής πληροφοριών για τις εταιρείες αυτές στις χώρες οι οποίες θα υποβάλουν σχετικό αίτημα. Επίσης τώρα ε, είναι δυνατόν η ανταλλαγή πληροφοριών για αυτές τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες πριν δεν ε, ήταν δυνατή διαδικασία ενώ τώρα έχει, γίνει, έχει καταστεί δυνατή. Όσον αφορά τους ε, beneficial owners, τους ε, πραγματικούς δικαιούχους πρέπει να σας πω ότι ήδη ο Παναμάς προσπαθεί να ενδυναμώσει τις ρυθμιστικές του αρχές. Έχουμε λοιπόν και μια ρυθμιστική αρχή η οποία ρυθμίζει μεταξύ άλλων τις ανώνυμες εταιρείες αλλά και άλλες μορφές επιχειρηματικές ε, οι οποίες ε, ε, δεν εκαλύπτονται μέχρι τώρα. Ε, οπωσδήποτε λοιπόν χρειάζεται η εξακρίβωση όλων των στοιχείων και ότι δηλαδή να εξακριβώσουμε ότι πράγματι εφαρμόζεται το νομοθετικό πλαίσιο αυτά μπορώ να σας πω, υπογραμμίζοντας για μία ακόμα φορά ότι ο Παναμάς ε, ε, είναι ε, πεπισμένος ότι ναι, είναι σημαντικό να υπάρχει νομοθεσία, να υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, ωστόσο αυτό δεν μπορεί από μόνο του να φέρει αποτελέσματα εάν δεν έχουμε και μία σωστή εφαρμογή και ε, εν πάση περιπτώσει, ε, εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν αποτελούν πρόκληση μόνο για τη δικιά μου χώρα. Είναι μια συνολική πρόκληση, αφορά το σύνολο ε, του, των χωρών. Ε, και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω και σας λέω και σας το υπογραμμίζω ότι αυτά που είπα εδώ και αυτά που κάνει η χώρα μου δεν είναι μονάχα λόγια. Προχωράμε και στην εξακρίβωση, προχωράμε και στην εφαρμογή. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Γκράντερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε κύριε Αντιπρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Πρεσβευτά. Άδικο θα ήταν η παρουσία της ε, Αντιπροέδρου να, ε, ε, να εξελιχθεί σαν να την είχαμε φέρει στην Επιτροπή των στοιχείων του Παναμά, των Panama Papers, αυτή τη διαρευνητική ε, επιτροπή. Θα ήταν άδικο, ειδικά για μας που γνωρίζουμε και αγαπάμε την ε, περιοχή αυτή του κόσμου. Και θα ήταν πραγματικά... Ε, είναι πραγματικά άδικο να γνωρίζει κανείς που δεν ξέρει ήδη τη χώρα, να γνωρίζει τον Παναμά μόνο μέσα από αυτά τα γρανάζια της Επιτροπής. Αυτό θα ήταν αδικία. Η χώρα σας είναι μεγάλη χώρα και πραγματικά έχει ιδιαίτερα σημαντική και ζηλευτή μπορώ να πω οικονομική ανάπτυξη. Ε, ε, επίσης όσον αφορά και το περιβάλλον είδαμε αυτό το μεγάλο έργο το οποίο ε, είχε, και πάρα πολλούς κινδύνους αυτό το μεγάλο έργο της, διόργας, της διάνοιξης μάλλον της διόργας που εφαρμόστηκε ήταν πάρα πολύ καλό. Έλεγα λοιπόν ότι εάν δούμε τον Παναμά μόνος με τα Panama Papers θα ήταν άδικο. Ωστόσο ε, είναι οι προκλήσεις πάρα πολύ μεγάλες. Εσείς είστε μια χώρα ε, που βλέπει και τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό. Ε, είσαστε μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει και αυτόν τον νέο απεικιοκρατισμό της Κίνας. Ε, και αποτελείται πραγματικά ένα σύμβολο ε, για την ανάπτυξη ε, νέων νομοθετικών και οικονομικών διασφαλίσεων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε το θέμα από πάρα πολύ κοντά. Η απάντησή σας, η ανταπόκριση του Παναμά ήταν άμεση και πραγματικά εσείς με διαφάνεια ε, και με ε, μεγάλη ενέργεια και θετική διάθεση ε, ξεκινήσατε την προσπάθεια. Τον προηγούμενο Σεπτέμβρη ο Παναμάς υπέγραψε την Συμφωνία για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης ο Παναμάς έχει δημιουργήσει πλέον νομοθεσία η οποία υποχρεώνει την καταχώρηση των εταιριών σε ένα μητρό επιχειρήσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλες, ε, ε, όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να δίνουν πληροφορίες ε, για την χώρα και για τις Εταιρείε οι οποίε ε, λειτουργούν εκεί. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Μπορεί να κάνουμε πάρα πολλέ αναλύσει και εδώ στο Κοινοβούλιο αρεσκόμαστε ιδιαίτερω ε, σε τέτοιου είδου ε, σε τέτοιου είδους αναλύσεις και έχουμε μάλιστα περισσότερο την τάση να κοιτάμε τους άλλους και να μην βλέπουμε και λίγο στις δικές μας χώρες και να μην βλέπουμε τα του οίκου μας πρώτα. Υπάρχουν βεβαίως και άλλα στοιχεία όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα που Μα απασχολούν πάρα πολύ και όταν κάνουμε συμφωνίε κτλ. Εν πάση περιπτώσει, η άποψή μου για τον ε, Παναμά σήμερα είναι πάρα πολύ θετική. Ε, η άποψή μου για τις προοπτικές που έχει ο Παναμάς είναι εξαίρετε. Υπάρχουν και άλλες χώρες ε, βεβαίως, αλλά πιστεύω ότι εσείς ειδικά θα πρέπει να είσαστε υπερήφανοι για τη χώρα σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Κράντε. Η κυρία Βέμπερ. Ah, Ευχαριστούμε πολύ. Καλώ ορίσατε κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για τι παρατηρήσει σα. Πρέπει να σα πω ότι εγώ συμφωνώ με τον Λίσαντα ε, ε, σχετικά με τη γνώμη που έχει για τον Παναμά. Αλλά έχω και μια ερώτηση η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο συμπληρωματική σε σχέση με την παρουσίασή σα. Στα πλαίσια τη ε, Eurolat εμεί δουλέψαμε πολλά χρόνια για να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να καταπολεμηθεί η διαφθορά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Λατινική Αμερική. Τι γίνεται με την χρηματοδότηση των ε, πολιτικών κομμάτων, των υποψηφίων στις εκλογές κτλ. Ε, αυτά τα διοικητικά νομοθετικά μέτρα ε, ε, που αναλαμβάνεται στον Παναμά θα έχουν κάποια επίπτωση στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών υποψηφίων σε εκλογές. Ευχαριστώ. Ναι. Ε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Φαρία. Εάν μπορείτε να κάνετε τι ερωτήσει σα πιο σύντομα, γιατί ο χρόνο μα πιέζει πάρα πολύ και για την κυρία Αντιπρόεδρο, αλλά γιατί θα πρέπει να φύγουν και οι διερμηνεί μα. Του οποίου ευχαριστώ ιδιαίτερα για την υπομονή που δείξανε και για το χρόνο που μα αφιερώσανε. Eh, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αντιπρόεδρο που ήρθε και να υποστηρίξω τα όσα είπε. Η χώρα σας είναι χώρα εταίρος, περιμένουμε πολλά βεβαίως. Κανείς δεν θέλει να καταδικάσει κανέναν και θα ήθελα να πω ότι ε, θα ήθελα να συγχαρώ τον πανόμα για την ε, ε, διεύρυνση της ε, διόρυγας, την οποία έχω ε, επισκεφθεί δύο φορές και έχω μείνει έκθαμβος από το μέγεθος του έργου. Βλέπουμε από τα όσα συστήσαμε μέχρι τώρα ότι έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες για την βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών ο Παναμάς με τις άλλες χώρες. Ξέρετε κύριε Πρόεδρε ότι Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις και από τη δική μου χώρα, εμπλεκόμενες στο σκάνδαλο του Παναμά. Θέλουμε να διερευνήσουμε τις υποθέσεις αυτές και, ξού, και διατυπώνω τις ερωτήσεις μου. Πώς μπορείτε να βελτιώσετε τη φήμη του Παναμά και πώς μπορείτε να βελτιώσετε την ε, εφαρμογή, να προχωρήσετε στην κύρωση και να προχωρήσετε στην εφαρμογή μετά της ε, Συμφωνίας για την Αμοιβαία Διοικητική και Φορολογική Συνεργασία και Αρρωγή. Και ιδιαίτερα οι τράπεζες στη χώρα σας. Ε, πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το, το φαινόμενο και τις δραστηριότητε τους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μιλάω γαλλικά. Δεν ξέρω, γιατί δεν έχω διερμηνία από τα γαλλικά, ε, εάν οι συνάδελφοι θα ε, έχουν ήδη διατυπώσει τις ερωτήσεις τους. Σας ενημερώνουμε ότι σε δύο λεπτά θα πρέπει να φύγουμε, δυστυχώς. Ε, έχουμε κράτη τα οποία ε, έχουν, ε, όπως ο Παναμάς, ακολουθήσει πρακτικές όχι θεμίτες. Έχετε αναπτύξει βέβαια μεγάλες προσπάθειες για τη διαφάνεια που το 2016 επιστεγάζονται με τη μαύρη λίστα του ΚΑΦΗ. Επίσης ε, προχωρεί ο Παναμάς στην κύρωση της Σύμβασης για την Αμοιβαία Διοικητική και Φορολογική Συνεργασία ε, για την ε, Επιτροπή Ειδικών λοιπόν που, δημοσιο... που δημοσίευσε μια έκθεση τον Νοέμβριο του 2016 ένα δημόσιο μητρό μετόχων ή ε, δικαιούχων δεν έγινε δεκτό ως λύση. Μπορείτε λοιπόν να μας εξηγήσετε αυτή την απόφαση και επίσης για την αμοιβαία αρρωγή στα φορολογικά θέματα πώς προχωρούν οι διμερείς συμφωνίες για την ανταλλαγή απόψεων και δυστυχώς τώρα θα πρέπει να σταματήσει η διερμηνία. Ευχαριστούμε και μίλησε το λόγο έχει η κυρία Αντιπρόεδρος. Muchísimas gracias eh, por las preguntas que me han sido formuladas, por los comentarios positivos hacia mi país, por el reconocimiento que han hecho a,